Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε. Έρχεται και ο κόσμος. Καλώς ορίσατε καταρχάς. Ξεκινούμε με μια ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σορίζω τους προσκεκλημένους μας. Τζένιφερ Κάστερ, Διευθύντρια του ειδικού προγράμματος του Ινστιτούτου Σίλη στην Πράγα, Αζού Κίπουλα, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, και Ελίζαμπετ Ντέβεκ, διευθύντριες προγράμματος του Διεθνούς Ινστιτούτου προσωρινή προσωρινής Βασική προϊότητα για την Επιτροπή μας, όπως αναφέρεται και στην ετήσια έκθεση που υιοθετήσαμε πέρσι στην Ολομέλεια, είναι η υποστήριξη των ε, υπερμάχων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε συζητήσει το θέμα της εφαρμογής των καθοδητήριων γραμμών της Ένωσης προς ε, όφελος των ε, υπερμάχων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, μεταξύ άλλων δικηγόρους κλπ. Η συνοχή του προγράμματος είναι ένα από τα βασικά θέματα που αναφέρονται στην πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό παραμένει πρόκληση και σε ό,τι αφορά τις, α, τις ε, απαντήσεις στις απειλές προς τους υπέρμαχους των δικαιωμάτων ανθρώπου. Η Ένωση έχει δεσμευθεί πολιτικά και έχει και έναν μηχανισμό χρηματοδότησης ειδικό. Μία απάντηση πολιτικής είναι να παρέχουμε προσωρινή προστασία και έκτακτη βοήθεια σε άτομα που, των οποίων η ζωή τους απειλείται στην πατρίδα τους. Ωστόσο, οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετωπίζουν ε, πολλά νομικά και πρακτικά εμπόδια όταν αναζητούν προσωρινή προστασία στην Ένωση, ιδίω για να πάρουν μια γρήγορη ε, βίζα για να μπουν στην Ένωση. Πρέπει να πούμε εξ αρχή ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να φύγουν από τη χώρα του ω το μέσο όταν οι διώξει και οι απειλέ εναντίον του είναι σοβαρέ και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση προσπαθούν να μείνουν κοντά στην πατρίδα τους, στην ίδια περιοχή. Όταν φεύγουν, συνήθως φεύγουν προσωρινά, προσπαθώντας να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι ένα θέμα που συχνά επίσης παρανοείται. Είναι σαφής ο στόχος να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς και να εντάξουμε προγράμματα δεν, δεν αρκεί όμως αυτό και δεν ανταποκρίνεται στην λογική και πρακτική των προξενικών αρχών των χωρών τη Ένωση. Έχουμε μεταξύ μας κάποιου ομιλητέ που θα υπογραμμίσουν τι προκλήσει, θα προτείνουν συστάσεις για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Ελπίζουμε ότι η σημερινή ανταλλαγή απόψεων θα διευκολύνει επίσης ε, παρόμοιες συζητήσει ε, και στις αντίστοιχες ομάδες εργασία του Συμβουλίου πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών εμπλέκονται επίσης στις σχετικές συζητήσεις. Τον Νοέμβριο πέρσι στην Πράγα μια σειρά μικιό συζήτησε το θέμα αυτό διατυπώνοντας συστάσεις για να αλλάξει το σύστημα θεωρήσεων για τους υπέρμαχους των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όπως σας είπα είχαμε, έχουμε δύο προσκεκλημένους ε, μαζί μας ε, στην, ε, από το Ινστιτούτο Σίλη στην Πράγα και θα μιλήσουμε για τις συστάσεις. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή μας, είναι τιμή μου να έρθω εδώ, που έχουμε εδώ, όχι μόνο ειδικό σε θέματα πολιτικής μετανάστευσης, αλλά ως ε, νομικός, με μια σειρά ιστοριών για να αλλάξουμε το την προοπτική για ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ένωση έχοντα διοκόμενοι διότι υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων στην πατρίδα τους. Πολλοί από αυτούς θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για σκοπούς που για μικρό χρονικό διάστημα προσπαθώντας να ενημερώσουν για την λαμπρή δουλειά που κάνουν. Η δουλειά μου, το έργο μου στην Πράγα είναι να παράσχω σε αυτούς τους ανθρώπους, ε, ακτιβιστές ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και άλλες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, για να τους βοηθήσω να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην περιοχή τους, δίνοντάς τους εύκολη πρόσβαση στην, ε, στις θεωρήσεις, κάτι που συχνά οδηγεί σε βελτίωση της πραγματικής κατάστασης. Ο στόχος μου είναι να διευκολύνουμε την κατάσταση στους πολίτες ε, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου ανά την Ένωση και να δούμε πώς επηρεάζει αυτό. Το συμπέρασμα είναι ότι τα προβλήματα αυτά είναι ευρύτερα, δεν είναι μόνο δική μου εμπειρία και από αυτό γεννήθηκε το έργο αυτό πολλές οργανώσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου έκαναν έρευνες, βοήθησαν ε, μια σειρά συστάσεων στην... Ε, Τώρα, για να είμαστε σαφείς, ε, εμείς υποστηρίζουμε συστάσεις για την πρακτική έκδοση θεωρήσεων βραχίας διαμονής ή 90 ημερών. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν υφιστάμενοι μηχανισμοί για προσωρινές θεωρήσεις ή προσωρινή μετακίνηση ατόμων που προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά αυτό δεν ήταν το κέντρο των ε, της προσοχής μας. Ε, η... Μεταξύ των ΜΚΟ και των ε, δομών πολιτικής πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος του περιορισμού του χώρου των ανθρώπων αυτών σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε, να, δημιουργήσουμε, να μας να δημιουργήσουμε ισχυρότερες σχέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό υποστηρίζεται από μια σειρά κρατικών και ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων. Η μείωση του ελεύθερου χώρου σημαίνει ότι πολύ συχνά οι πολίτες αυτοί πρέπει να μπορέσουν να γίνουν κάτι πιο ευέλικτο και να παράσχουν το δικαίωμα, ουσιαστικό δικαίωμα προστασίας τους όταν ε, στην ε, κοινωνία της χώρας ε, προέλευσής τους δεν μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Η έκθεση, αντίγραφα των οποίων υπάρχουν και στην αίθουσα, συνδυάζει την ανάλυση και την έρευνα για την πολιτική θεωρήσεων της Ένωσης και τους σχετικούς μηχανισμούς με ανώνυμες σε 120 ατόμων από 10 χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση και τη Τουρκία. Το εντοπίζει τη, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων ανθρώπου όταν ζητούν θεωρήσει για να έρθουν στην Ευρώπη. Οι συνάδελφοί μα στι μεγάλε οργανώσει προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό σαν δικό του εργαλείο διαμόρφωση πολιτική όταν κάνουν λόμπι σε εθνικό επίπεδο. Να τομίσω κάποια από τα στοιχεία της έρευνας που θεωρούμε σημαντικά και που βεβαιώνουν κάποιες από τις εικασίες μας για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Όπως σας είπα, κάναμε έρευνα σε 10 χώρες για να καταλάβουμε δημογραφικά, δημογραφικά μοντέλα. 23% 23% είναι γυναίκες, 11% ε, από την κοινότητα LGBT. νέοι, οι περισσότεροι ήταν νέοι ακτιβιστές ή νέοι επαγγελματίες. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν κερδίζουν πολλά χρήματα, αγωνίζονται για τα προστοζήν και 53% από αυτούς ε, κερδίζουν λιγότερο από 5.000 ευρώ το χρόνο. Ταξιδεύουν συχνά στην Ένωση, 35% από αυτούς ε, έχουν, ταξιδεύουν πάνω από 5 φορές το χρόνο δεν έχουν η πλειοψηφία τους visa Σέγγεν. 20% έχουν πάνω από 5 θεωρήσεις Σέγγεν στο διαβατήριό τους. Η λογική, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η λογική της έκδοσης θεωρήσεων είναι για συγκεκριμένες δραστηριότητε. Για να πάει ας πούμε σε μια, σε μια διάσκεψη, η συνάδελφος θα μιλήσει για τα θέματα αυτά. Ωστόσο οι πρακτικές αυτές ε, ε, συχνά σημαίνει ότι οι θεωρήσεις τους δίνεται από πολλά κράτη-μέλη, διαφορετικά κράτη-μέλη, με ε, καθυστέρηση και επανειλημμένη ε, πληρωμή του κόστου στη θεωρήσεως. Πολλοί από αυτούς δεν ε, ε καταφέρνουν να κάνουν το έργο αυτό μόνο, μόνοι τους και συχνά παίρνουν υποστήριξη από τρίτους. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις ε, είναι η εξή 66% ο χρόνος για τις θεωρήσεις και για την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων είναι υπερβολικά μεγάλος. 65% μίλησαν, ε, είπαν ότι, ότι το κόστος ήταν πολύ μεγάλο και 22% εξέφρασαν ε, ταπείν, αισθάνθηκαν ταπείνωση κατά τη διαδικασία αυτή. Πολλοί από αυτούς τόνισαν ότι δεν μπορούσαν να παράσχουν πιστοποιητικά τραπεζικά για να πείσουν τα προξενία ότι έχουν ε, ότι έχουν την οικονομική υποστήριξη για να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς χρειάζεται να ζητήσουν δάνειο από φίλους, από οικογένειες μόνο και μόνο ή να βάλουν χρήματα στο λογαριασμό τους για να δείξουν ότι έχουν χρήματα στις τράπεζες. Το οικογενειακό στάτους, ε, το, καθεστώς, ε, το οικογενειακό καθεστώς είναι πολύ σημαντικό σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές, ιδίως για, τους, ε, για την κοινότητα LGBT, όπου συχνά αισθάνονται ότι αν δεν αναφέρουν οικογένεια μπορεί να κινδυνεύσουν να μην λάβουν αυτή την θεώρηση. Η κοινότητα αυτή στην πράξη, επειδή χρειάζεται να φύγει πολύ συχνά, δεν μπορεί να βρει μόνιμη δουλειά. Οι περισσότεροι από αυτού είναι freelance, είναι, δεν έχουν σταθερό επάγγελμα, κάτι που ισχύει, στην ουσία μετράει ει βάρο του όταν ζητάνε βίζα. Να επανέλθω στο θέμα τη κινητικότητα και να τονίσω πόσο σημαντικό είναι και πόσο κρίσιμο είναι για αυτή την κοινότητα των ανθρώπων. Η πίωση στους ακτιβιστέ αυτέ τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά με μεγάλη αύξηση των πιέσεων σε ακτιβιστές τις χώρες τη περιφέρειας της Ευρώπη. Μια ανοιχτή θεώρηση Σέγγεν είναι βασικό εργαλείο για πολλούς τέτοιους ανθρώπους, όχι μια πολυτέλεια για λίγους. Θέλω να τονίσω επίσης ότι αυτό είναι μια κοινότητα που θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα της. Όπως λέει και το Frontline, θέλουν να γυρίσουν στην Ευρώπη για την ευημερία, για επαγγελματική ανάπτυξη και για δικτύωση πριν γυρίσουν να ξαναπαλέψουν στην πατρίδα τους. Δεν, δεν για αυτούς, ε, δεν, δεν που αρρωγεί να τους δώσει κανείς βίζα. Είναι ένα κομμάτι, το θεωρούν ένα κομμάτι της ταλαιπωρίας τους, αλλά εμείς πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Στις συστάσεις που δίνουμε θα δείτε και κάποιες συστάσεις για το τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν την κατάσταση. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συνεπείς προσπάθειες εναρμόνισης των εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών είναι βασική παράμετρος. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ριζικές νομοθετικές αλλαγές. Η πρώτη σύσταση λοιπόν είναι να υπάρξει μία ειδική γλώσσα για τους υπέρμαχους των δικαιωμάτων ανθρώπου στο εγχειρίδιο θεωρήσεων Σέγγεν, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέλη της οικογένειάς τους και την και να, ε, χωρίς, να, ε, να λαμβάνουν υπόψη τις παράμετρους που συχνά χρησιμοποιούμε. Έσοδα, εισοδήματα, οικογένεια κλπ. Σε ό,τι αφορά την χρήση τώρα του συστήματος αυτού, ε, πρέπει να μπορούμε να παράσχουμε στοιχεία επαρκή για την έκδοση θεωρήσεων για τα άτομα αυτά. Να πω δύο λόγια ευχαριστειών τώρα στην Αναλύσα Αναλώνη πρώτα, καθηγήτρια στο Λονδίνο, που έδωσε το νομικό πλαίσιο της έκθεσής μας στους συναδέλφους από το Ινστιτούτο Σίλη που μας βοήθησαν να κάνουμε την έκδοση και τον ε, συνάδελφο που μας βοήθησε να κάνουμε την ε, συλλογή των δεδομένων. Να ευχαριστήσω και όλους σας για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσουμε τις ε, απόψεις αυτές. Με μικρές αλλαγές θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην αντιμετώπιση των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την παροχή, ε, εύκολη, την ευκολότερη παροχή βίζα στους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε. To Arzu Gaybula, who is a journalist and activist from Azerbaijan. Her testimony is relevant to us not only as someone who was forced to leave her country because of threats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 Και έτσι εξηγήθηκε από αυτού που με κάλεσαν ότι πρόκειται να καλυφθούν τα έξοδα και δεν χρειαζόταν επιπλέον δικαιολογία, δικαιολόγηση των χρημάτων που είχα στην τράπεζα. Αλλά ο υπάλληλο ανησυχούσε και μου έλεγε ότι θα έχει πρόβλημα εάν του δώσω το συγκεκριμένο δικαιολογητικό και το κέντρο έκδοσης θα είχε πρόβλημα γιατί θα ήταν ημιτελής η αίτηση, ελλειπής. Οπότε πήγα στην τράπεζα, ευτυχώ είχε ένα υποκατάστημα, πήγα, περίμενα άλλη μια ώρα γιατί δεν ήταν εκεί ο υπάλληλος που χρειαζόταν, που έπρεπε να υπογράψει και μετά έπρεπε να επιστρέψω στο κέντρο έκδοσης ε, ε, όμως ε, είχαν διάλειμμα μεσημεριανό, έπρεπε να περιμένω άλλη μια ώρα και μετά άλλη μισή ώρα γιατί μετά είχαν έρθει άλλοι που προηγούντο. Απλώς για αυτό το ένα δικαιολογητικό που δεν χρειαζόταν καν για τη συγκεκριμένη βίζα. Και πήρα την τριμηνία και όταν γύρισα από το πανεπιστήμιο θα πρέπει να κλείσω ένα ραντεβού πάλι γιατί έπρεπε Είχαμε ένα φεστιβάλ, κάτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, γύριζαν μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ και εγώ έπρεπε να εμφανιστώ εκεί. Τέλος πάντων. Άρα η εμπειρία μου με το κέντρο έκδοσης θεωρήσεων ήταν έτσι. Όταν έλεγα στον υπάλληλο ότι δεν χρειάζομαι δικαιολογικό, έλεγε όχι, πρέπει να το υποβάλλετε. Και ε, έκαναν μηχανικά τη δουλειά τους δεν του ένοιαζε <clears throat> ό,τι εξηγούσε ποιο είσαι, τι κάνει, χρειάζεσαι, δεν χρειάζεσαι το δικαιολογητικό. Βέβαια εντάξει, σε μεταχειρίζονται καλύτερα όταν πληρώνει κάτι έξτρα. Όταν πας ε, στο γραφείο αυτό, έχουν ε, ωραίου καναπέδες, πολυθρόνε, σοκολατάκια, καφέ. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν οι κοινοί θνητοί Ε, επίσης επανειλημμένα, έκανα αιτήσει, επανειλημμένα πλήρωσα και... Κοίταξα να δω πόσε είναι οι βίζε που έχω πάρει αυτά τα χρόνια. Μία εξάμηνη, τρει τετράμινε, δύο αιτήσει. Τελευταία, τελευταία ήταν ενό έτους και έτσι γλίτωσα, γλίτωσα σωρό έξοδα τα τέλη του κέντρου, τον ΦΠΑ, το τακτικό τέλος και όταν άρχισα να σας μιλώ σήμερα σας είπα ότι θεωρώ πως είμαι τυχερή γιατί να ας πούμε έχω έναν φίλο πρώην πολιτικό κρατούμενο αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο πέρσι και έγινε κατά την πολιτική κρατούμενη και όλη η οικογένεια είναι Κάνανε μια αίτηση για να ταξιδέψουν στην Γερμανία για κάποια εκδήλωση και τους είπαν όχι. Και δεν ε, τους το εξήγησαν, είπαν κάποια δικαιολογία. Και είπε ότι ήταν ταπεινωτικό ο, αυτός ο φίλος πιο ταπεινωτική αυτή η απάντηση γιατί έχω κάνει πέντε χρόνια φυλακή και ήθελα να μεταναστεύσω μετά από τόσα χρόνια. Δεν θέλω να περάσω τη ζωή μου στη φυλακή. Να, άλλο ένα παράδειγμα τελευταίο. Άλλος φίλος και αυτός δημοσιογράφος που είχε κάποια προβλήματα υγείας αυτή η κοπέλα είχε ε, κάποια επέμβαση για ένα τμήμα της λεκάνης και επί έξι χρόνια δεν μπορούσε να πάει για την θεραπεία της, για την αγωγή της, γιατί της είχαν μπλοκάρει τη βίζα, είχε μπλοκαριστεί στη χώρα της, ε, ήταν σε εξορία, ήταν αυτή σε κάποια μαύρη λίστα, λόγω του που δούλευαν, σε ποιον οργανισμό δούλευαν. Και υπήρχε ε, μια έρευνα εις βάρος και με αντικείμενα αυτό τον εκδοτικό οργανισμό που δούλευε. Άρα τη είπανε όχι για βίζα. Δεν μπορεί να γυρίσει. Είπαν και σε αυτή ανήπαντρε. Δεν είχε ε, αρκετά χρήματα στην τράπεζα να αποδείξει ότι μπορεί να ζήσει με αυτά. Και, και ασχολήθηκε με πήγε σε διάφορου οργανισμού, χωρί σύνορα και άλλου. Τη δώσανε κάποιε συστατικέ επιστολέ, ε, αλλά δεν απέδωσαν. Άρα θα έπρεπε τελικά να, να μπούμε πειρατικά στο σύστημα και οπότε με άλλα κανάλια να φτάσουμε ε, στο... και επίσης υπήρχε, κάναμε επαφή και με κάποιον Αμερικανό γιατρό για να βοηθήσει να δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε κύριε Γκίμπουλα. Όταν άκουγα την παρουσίασή σα, σκέφτηκα ότι αυτό είναι το μέλλον και για του κατοίκου τη δική μου τη χώρα. Τέλο πάντων, αστείο ήταν αυτό μια προσωπική μαρτυρία πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι πολλοί ακτιβιστέ που ασχολούνται με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δίκτυο για ε, τι πόλει των ε, μεταναστών ICON, που είναι μέλο τη πλατφόρμα επανακατάσταση. Ε, εδώ έχουμε την κυρία και την προ... τη διευθύντρια, που θα μα δώσει τη δική του προοπτική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, μέλη της Υποεπιτροπής, κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ εκ μέρους της ICON, ε, του Διεθνούς Δικτύου των ε, Πόλεων για Μετανάστες. Να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Είμαστε μια, ένας οργανισμός με ανεξάρτητα μέλη που θέλουμε να ενισχύσουμε ε, τους μετανάστες διεθνώς. Έχουμε καμιά εβδομενταριά μέλη, ε, όπου συμμετέχουν πόλεις με κυβερνητικές οργανώσεις και πανεπιστήμια. Κάθε πόλη προσφέρει για δύο χρόνια ε, κατοικία ε, σε δημοσιογράφους, συντάκτες άρθρων ή καλλιτέχνες που διώκονται. Είναι προσωρινή η στέγασή τους. Είναι για ανθρώπους που δεν μπορούν πλέον να εργαστούν ελεύθερα στις χώρες τους. Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλλιτέχνες που πολλές φορές ε, ε, πρέπει να υποστούν διακριτική μεταχείριση λόγω της έρευνας ή των αφηγημάτων που γράφουν ή των άρθρων τους και δεν μπορούν πλέον να εργαστούν από το σπίτι τους. Από τις 70 πόλεις, περίπου 65, βρίσκονται σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπόλοιπε στην Αμερικανική Ήπειρο. Θέλω να μιλήσω και ως μέλος της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσωρινή μετακατάσταση. Ε, μιλάμε για, για μια πλατφόρμα για διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την προσωρινή ε, μετακατάσταση των ε, προσπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος είναι να διευκολύνει τη συνεργασία και το συντονισμό των παραγόντων που ασχολούνται με την προσωρινή μετακατάσταση των προσπιστών, των ακτιβιστών. Η πλατφόρμα είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάπτυξη και ο συντονισμός της πλατφόρμας βρίσκεται στα χέρια ε, του Protect Defenders EU, ένα μηχανισμό για την προστασία των ακτιβιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε περίπου 50 αυτή τη στιγμή ως μέλη και τα δύο τρίτα ε, βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάθε κάτω μέλο πρέπει να προσφέρει ιδέε για μέτρα για σαφή ε, προστασία και γρήγορη προστασία ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτε χώρε. Όπου χρειάζεται δηλαδή να δοθούν κατεπηγόντω θεωρήσει ή να διευκολυνθεί η ε, άμεση ε, προσφορά στέγη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσωρινή μετεγκατάσταση τώρα. Κατά την άποψή μου, αφορά ε, τρεις περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα είναι μια επίγουσα ανάγκη για να ξεφύγει κανείς από κίνδυνο ή κάτι που συμβαίνει εκτάκτως. σε άλλες περιπτώσεις είναι σχεδιασμένη, προγραμματισμένη μια προσωρινή μετακατάσταση τριών μηνών που σκοπό έχει να έχει μια ανάπαυλα ο υπέρμαχος ε, να ξεκουραστεί ή να βελτιώσει το δίκτυό του ή να μπορέσει να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο σκοπό ή μπορεί να είναι ένα προσωρινό μέτρο που προέρχεται από τις σοβαρές απειλές που μπορεί να έχει δεκτεί κάποιος υπερμαχός από ε, απειλές φυλάκισης, παρενόχληση, ε, σωματικές βλάβες και ούτω καθεξής. Η θεώρηση Σέγγεν είναι συνήθω 90 ημέρε. Συζητάμε με διάφορε εθνικέ κυβερνήσει και μεταναστευτικέ αρχέ σε χώρε όπου ε, συμμετέχουν στο δίκτυό μας για να δούμε αν μπορεί το διάστημα αυτό να αλλάξει. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι μπορούμε να κάνουμε. Στη Δανία, όταν μιλήσαμε με τις αρχές μετανάστευσης, δεν βρήκαν καμία δυνατότητα στην υπάρχουσα νομοθεσία για να αλλάξει η άδεια παραμονής. Έτσι, με τις δανέζικες αρχές και το ε, Συμβούλιο Καλλιτεχνών ε, του, της Δανίας ε, ασκήσαμε πίεση για να αλλάξει νομοθεσία. Η, Βουλή της Δανίας άρναξε τον νόμο για τη μετανάστευση, οπότε επιτρέπεται σε καλλιτέχνες που προσκαλούνται σε μια πόλη μέλος της, του Διεθνούς Οργανισμού να πάρουν διετία διαπεραμονής μαζί με τις οικογένειές τους. Υπάρχει και περιορισμένη άδεια εργασία που επιτρέπει να εργαστούν αλλά στον επαγγελματικό του κλάδο. Τα μέλη τη οικογένεια παίρνουν επίση άδεια παραμονή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό τη Σουηδία. Η, Σουηδι... η Σουηδική κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δουλειά μα. Και αυτό λόγω τη άσκηση πίεση ε, των πόλεων που βρίσκονται στη Σουηδία και είναι μέλη του δικτύου μα. 25 αυτή τη στιγμή. Έτσι το ΑΕΚΟΝ, το Σουηδικό Συμβούλιο Καλλιτεχνών και η Μεταναστευτική Αρχή, μάλλον προσέγγισαν τη Μεταναστευτική Αρχή της Σουηδίας για να δουν τι μπορεί να γίνει με τη θεώρηση και την άδεια παραμονής για καλλιτέχνες και δημοσιογράφους και αν μπορούν να μείνουν στη χώρα ε, ως δύο χρόνια. Η μεταναστευτική αρχή είπε ότι εφόσον οι επαγγελματίες μπορούν να κερδίζουν τη ζωή τους, μπορούν να ετηθούν ε, άδειε, που ε, χορηγείται σε αυτούς που λέγονται αυτούς που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίε. Σε αυτούς που εργάζονται ως ελεύθεροι Έτσι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνε και ε, συγγραφείς που προσκαλούνται στη Σουηδία μπορούν να κάνουν αίτηση για διετή άδεια. Η ΑΕΚΟΝ βεβαίως ε, η ICON ελέγχει κατά πόσο τα στοιχεία του κάθε καλλιτέχνη δημοσιογράφου, ε, συγγραφέα, συντάκτη άρθρων ή ακτιβιστή ε, είναι σωστά. Επίσης, μπορεί να ε, αιτηθεί ο άνθρωπος αυτός μόνιμη άδεια παραμονή στη Σουηδία, εφόσον μπορεί να κερδίσει τη ζωή του. Υπάρχει και γι' αυτό ειδικό έντυπο. Η πλειοψηφία όσων έρχονται σε εμά δεν θέλουν να πάρουν το καθεστώ πρόσφυγα. Θέλουν προσωρινώ να μετεγκατασταθούν για να μπορούν παρόλα αυτά να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσή του όταν θέλουν, να παραμείνουν σε επαφή με το κοινό του, τι εκλογικέ του περιφέρειε, τι κοινότητε του πληθυσμού τι οποίε προέρχονται για να συνεχίσουν να εργάζονται ω ακτιβιστέ. Σε άλλε χώρε όπου έχουμε μέλη ω Πόλη ως μέλη, έχουμε συνεργαστεί με μεταναστευτικέ αρχέ για να βρούμε λύσει και για να δούμε αν μπορούν οι άνθρωποι που προσκαλούνται να μείνουν ένα ω δύο χρόνια ε, στη χώρα με την προπόθεση να κερδίζουν τη ζωή του και επίση να μπορούν να επιστρέφουν στη χώρα προέλευσή του, Μαζί με τι οικογένειε του, που πρέπει να ταξιδεύουν με του ακτιβιστέ, αν και υπάρχουν πολλέ χώρε όπου αντιμετωπίζουμε δυσκολίε. Organizations who are member of the temporary relocation platform. Για την πλατφόρμα τώρα. Έχουμε παρόμοιε καλέ εμπειρίε από τη συνεργασία μα με τι εθνικέ μεταναστευτικέ αρχέ. Ιδίω όταν υπάρχει στήριξη από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων ή άλλου, δηλαδή την κυβέρνηση. Όπω το πρόγραμμα προστασία στην Ολλανδία που προσφέρει τρίμηνη άδεια παραμονή σε ακτιβιστέ και το Ίδρυμα του Αμβούργου για τους ε, πολιτικούς διοκόμενους που προσφέρει διετή άδεια παραμονή στη Γερμανία. Θα θέλαμε όμως περισσότερα κάτι μέλη να ε, υπερασπίζονται αυτές τις εναλλακτικέ για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυβερνήσει θα πρέπει να σκεφτούν το σύστημα θεωρήσεων μια προσωρινή άδεια παραμονή. Και θα έλεγα το εξή. Συνεργαστείτε μαζί μας με το ICON, ε, με, με τα μέλη της πλατφόρμα, γιατί εθνικός και περιφερειακός μπορούμε να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τους ε, ε, ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τις κυβερνήσεις και να βρουν τις κατάλληλες οργανώσεις για να τους ε, στηρίξει. Και όπου χρειάζεται να γίνουν και απαραίτητες προσαρμογές στην νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ντιβίκ. Οι συνάδελφοι 18 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, άρα πολύ χρόνο. Να σας ευχαριστήσω μόνο για όσα μας είπατε. Δεν είναι πάντα εύκολο, όπως είπατε. Αυτά που περιγράψετε για τη δική σας περίπτωση, για τη θεώρησή σας, Ελπίζω να μην συμβεί αυτό για τη Βρετανία, αλλά πρέπει να πω ότι όταν σας άκουσα σκεφτόμουν τι διοικητικά πράγματα πρέπει να κάνουμε για άλλα πράγματα. Πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό βάρος για όλους μας. Θα θέλαμε να ήταν ευκολότερα τα προβλήματά σας και για σας και για όλους. Αλλά Δεν ξέρω αν είναι ευκολότερο μόνο για όσους αγωνίζονται για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε σχέση με άλλους, αλλά πάντα, πάντως δεν είναι εύκολα. Και έχουν και την πίεση από πάνω. Νομίζω ότι Πρέπει να το δούμε το θέμα. Ευχαριστώ. Για τη δουλειά και για ό,τι κάνετε. Anybody from S&D who wants to raise anything? I pass the floor to Phil, please. Phil. Θα ήταν χρήσιμο να βρούμε έναν ε, γενικά αποδεκτό ορισμό γιατί μπείτε στη θέση του γραφειοκράτη που επεξεργάζεται τις αιτήσει. Τι θα πει υπέρμαχος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο ίδιος το λέει. Εγώ είμαι υπέρμαχος, άρα ο καθένας. Ή είναι κάποιος που τον λέμε εμείς. Μπορούμε να δούμε ας πούμε ένα μητρό που θα μπορούσε να δεχθούν οι αρχές. Έστω και αν αυτό πρέπει να το αναθεωρούμε. Δεν γίνεσαι δηλαδή ισόβια υπέρμαχος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το δούμε αυτό. Επίσης, Πρέπει να σας πω ότι το καθεστώς του Σέγγεν για τις θεωρήσεις είναι καλύτερο από το αγγλικό, από το βρετανικό. Εγώ είμαι αντιπρόεδρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Διεθνή των Φιλελευθέρων και έχουμε 22 μέλη. Ούτε ένας δεν είναι από την ίδια. Δύο, κάθε ένας είναι από άλλη χώρα. Το τι πρέπει να κάνουμε για να οργανώσουμε μια συνάντηση δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Επίσης, συνεργαζόμαστε με πολιτικούς, μεγάλους πολιτικούς. Τα γραφεία μας είναι στο Λονδίνο. Και πάλι δεν μπορούσαμε να βγάλουμε βίζα για τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Κονγκό για να έρθει στο Λονδίνο. Άρα χρειάστηκε να πάμε στο Παρίσι για να κάνουμε τη συνάντηση. Τέτοια είναι τα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζουμε. Άλλε φορέ κάποιο παίρνει βρετανική βίζα, αλλά όχι βίζα Σέγγεν. Είναι παράλογα τα πράγματα. Εμεί είμαστε πολιτική οργάνωση, αλλά έχουμε και καθεστώ μη κυβερνητικό οργανισμού. Είμαστε στο Συμβούλιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γενέβη και πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα μιλήσει, γιατί πρέπει να, αποφασι... πρέπει να μάθουμε ποιο θα καταφέρει να μπει στην Ελβετία. Και συνεχώ μιλάνε οι Ευρωπαίοι γιατί μπορεί να πάνε, ενώ δεν μπορεί να έρθουν οι Αφρικανοί. Άρα χρειαζόμαστε κάποια μορφή μητρώου πολιτικές προσωπικότητες και αγωνιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εγώ πρέπει να φέρω τώρα τον κύριο Κάμπτο από το Καμερούν τώρα για να μπορέσει να μιλήσει με την κυβέρνηση. Έφτασε στο Παρίσι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να... Δεν ξέρει ακόμα αν θα πάει στην Βρετανία. Δεν, δεν παρά, είναι παράλογη όλη η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη και χρειάζεται βέβαια να υπάρξει πρόοδος. Ευχαριστώ Φιλ. Χάνελ. Ένα πράγμα επί του οποίου μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι είναι το σύστημα θεωρήσεων που έχουμε δεν είναι το καλύτερο. Άσε που και οι Βρετανοί δεν χρειάζεται να είχαν δικό τους, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα. Η κατάσταση των αγωνιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι χειρότερη και διαφορετική. Αυτό κατάλαβα από τις συζητήσεις. Ε, μπορώ να φανταστώ ότι αν σου ζητούν, ας πούμε, τι έγινε, να, την, αν σου ζητούν να δείξεις ε, αντίγραφο του λογαριασμού, των κινήσεων του λογαριασμού στο τελευταίο τετράμινο, και αυτό φτάσει στους... Ε, τέλο πάντων στι αρχέ, μπορούν να δουν πού παίρνει τα λεφτά, να σε κυνηγήσουν στο δίκτυο ή να σε φέρνουν μπρο πίσω για να παίρνει βεβαιώσει κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα, να σου δώσουν βραχία διάρκεια θεώρηση. Ενώ είσαι ήδη μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κακή κατάσταση λοιπόν. και πραγματικά είναι πολύ προβληματικό. Να σας πω γιατί. Υπάρχει, είπατε ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Επιτροπή. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα της Ένωσης για αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τους καλούμε σε συναντήσεις για να βελτιώσουμε την κατάστασή τους και αν, αυτοί καλέ, και αν αυτά τα προγράμματα καλέσουν αγωνιστές να έρθουν, οι άνθρωποι δεν παίρνουν θεώρηση. Αυτή είναι η κατάσταση. Ασυνέπεια. Ό,τι πιο ασυνέπεια μπορεί να φανταστεί. Έρχεται, ξέρω εγώ, η Διεθνή Αμνηστία, η Greenpeace, το Frontline Defenders σε μία συνάντηση. Δείχνει ότι εμείς αναγνωρίζουμε ως αγωνιστή. Δηλαδή, άμα δεν είναι το θέμα να είναι ιστοδυναικές αγωνιστές. Όταν έρχονται σε ένα, όταν έρχονται για ένα συνέδριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ε, αγωνιστές για τα δικαιώματα του ανθρώπου θα είναι. Τι θα είναι. about the protection of human rights defenders. Έρχονται από χώρε που έχουν δύσκολη κατάσταση και τους βάζουμε και ακόμη περισσότερες δυσκολίες. Μ' αρέσουν οι συστάσεις, είναι συγκεκριμένες και λένε κατά βάση δείτε το εγχειρίδιο Σέγγεν και διδάξτε αυτούς που κάνουν τη διαδικασία. Και προτείνω να κάνουμε και μια άλλη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό με τους συναδέλφους στη ΛΥΜΠΕ που έχουν την εμπειρογνωμοσύνη για να υπάρχει μια συνεκτικότητα σε όλα αυτά. Γιατί αυτό είναι κάτι που μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα μεθυμίζω ότι έχουμε και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ. Εμείς παντού τους καλήσαμε. καλέσαμε. Άντε, να τους ξανακαλέσουμε, ίσως. Ε, η επόμενη, η κυρία Στρίξ, ε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, κοινή πρωτοβουλία είναι αυτή ε, τη δική μα Επιτροπή και τη ΛΥΜΠΕ. Εγώ ευτυχώ είμαι και στι δύο επιτροπέ και αυτό κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, γιατί έτσι ξεκαθαρίζεται το ότι η ευελιξία χρειάζεται πάρα πολύ, αλλά και η κινητικότητα, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να κινηθεί, να δουλέψει σε όλη την Ευρώπη, ε, οπότε θα θέλει κανείς ή χρειάζεται, χρειάζεται άμεσα να ε, το διεκπεριώσει και να φτιάξει το δίκτυό του και όχι πάντα με προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Οπότε καταλαβαίνω ποιο είναι το δίλημα όσον αφορά αυτό το κώδικα. Ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν. Μας είπατε επίσης ε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος της εγκατάστασης ε, και αυτό είναι διαβόητη, πολύ γνωστή δικαιολογία για απόρριψη. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Τα είπε και η Χάνα ότι υπάρχουν ε, και πολιτικοί λόγοι. Δεν θέλουν δηλαδή να κάποιες χώρες, από εκεί που έρχεται δηλαδή ο ετών, να, τις χώρες αυτές προέλευσης να τις ε, προσβάλλουν. Είπαμε, ε, μήπως θα πρέπει να διευρυνθεί ο ορισμό του ακτιβιστή. Συμφωνώ 100% αλλά έτσι είναι πιο μπερδεμένο. Τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη, τι ορισμό θα υιοθετήσουν και κατάλαβα τελευταίο μιλήτριο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουν ε, τα κράτη ότι συνεργάζονται και οι οργανισμοί ανθρώποι δικαιωμάτων ότι συνεργάζονται με κάποιον που είναι ακτιβιστής. Υπάρχει τέλος πάντων αυτό το περιθώριο στον κώδικα και θα πρέπει να γίνει ομοιόμορφη εφαρμογή από αυτή τη δυνατότητα που παρέχεται. να εκμεταλλευτούμε όλα τα περιθώρια που υπάρχουν για να υπάρχει αιτήσια διαιτήση σε βίζα πέραν του κώδικα. Οπότε να έχουμε συγκεκριμένα μια ρύθμιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μακροπρόθεσμη, να μην είναι ισόβια, αλλά να είναι δυνατόν έτσι να παρασχεθεί στους ακτιβιστές ε, κάποια διευκόλυνση, να μπορούμε να έχουμε πανευρωπαϊκή συνεργασία σε όλη την Ευρώπη. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Α, και κάτι πάρα πολύ σύντομα να σας πω. Νομίζω ότι πέραν των όσων ήδη ακούσαμε είναι και θέμα πολιτικό. Ένα μήνυμα ότι ε, αν ε, παίρνουμε στα σοβαρά την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές ως Ευρώπη να στείλουμε αυτό το πολιτικό ε, μήνυμα. Δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τους ακτιβιστές, θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε. Symbolic, very, ε, ε, um, Και πάρα πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε όλα αυτά να τα μεταρρυθμίσουμε, να τα τροποποιήσουμε. Ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Ποιος θα ήθελε τώρα να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ποια θα ήθελε πρώτη να απαντήσει. Um, I'd like Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το θέμα του Μητρώου θα με απασχολήσει γιατί εδώ υπάρχουν κάποια σημαντικά σημεία. Ποιος δίνει τον ορισμό γιατί πολλές φορές κάποιος που αυτοκαθορίζεται αρχίζει την επαφή με το προξενείο και έχουμε όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ε, ποιος είναι που δουλεύει αυτό το πρόσωπο και αυτό σας τονίζω. Δεν μιλάμε για πλήθη που προσέρχονται στο προξενείο και θέλουν να ε, ισχυριστούν ότι είναι ακτιβιστές. Θα ήταν επικίνδυνο. Θα πρέπει να ε, έχει φυσικά το περιθώριο να πει όχι, να απορρίψει την αίτηση ο υπάλληλος αλλά πρέπει να μελετήσει τα δικαιολογητικά, να το δει με άλλο μάτι. Ε, δεν νομίζω ότι γι' αυτό απαιτείται μητρό. Από την άλλη μεριά βέβαια το μητρό παρέχει ασφάλεια. Και όμως οι λίστες και τα στοιχεία διαραίουν. Πάνε αλλού. Οπότε αυτό είναι ρίσκο για τους σχετικούς συναδέλφους. Δεν ξέρω, τα ξέρουν καλύτερα εδώ οι παρακαθήμενες. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, λέει κύριε Αντιβίκ. Είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα πρέπει να έχουμε έναν ενιαίο κώδικα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σέγγεν. Αλλά δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε να γίνουν όλες οι διαδικασίες. Ό,τι είναι το πιο γρήγορο είναι και καλύτερη λύση. Κάθε κάτω μέλος πρέπει να δει τι θα κάνει. Ίσως να εργαστούμε με τον κώδικα των θεωρήσεων που έχουμε για να δούμε τι μπορεί εκεί να βελτιωθεί. Όταν ας πούμε κάποιος εγκριθεί μια πρώτη φορά, μήπως ε, να εγκρίνεται πιο εύκολα τη δεύτερη, χωρίς να πρέπει να τα ξαναφέρνει όλα τα δικαιολογητικά κάθε 6 μήνες. Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω πώς θα γίνει πιο απλό, πιο απλή διαδικασία. Αντί να έχω 15-20 θεωρήσεις στο διαβατήριο, νομίζω ότι κάποια στιγμή έχω αποδείξει ποια είμαι. Δεν σκοπεύω να έρθω και να μείνω σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο πράγματα τώρα για τους ορισμούς. Πώς θα γίνει ο ορισμός των υπερμάχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακτιβιστών. Είναι σαν να προσπαθούμε να ορίσουμε του πολιτικού κρατουμένου και αυτό μου θυμίζει πολύ και τα όσα έλεγε η κυβέρνησή μου, που έλεγε ότι δεν υπάρχει ένα ορισμό για του πολιτικού κρατουμένου. Οι 100 και πάνω που βρίσκονται στη φυλακή λοιπόν δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι παρόλο που είναι. Να, που είναι το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να υπάρχει ένα ορισμό που να καλύπτει όλα. Βάσει των προηγούμενων αναπηρίο μα τουλάχιστον. Τώρα για τα τραπεζικά στοιχεία. Σωστά το αναφέρετε. Διότι αν έχει παγώσει ο τραπεζικό σα λογαριασμό από την κυβέρνηση, αυτή που δεν σα αφήνει να φύγετε, τι να γίνει τότε. Δεν μπορεί να δείξει ούτε τα στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων μηνών, αφού ήταν στοιχεία παγωμένα. Θα πάψω εδώ. Δύο λεπτά έμειναν. Μια χαρά. Νομίζω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Home, έχουμε εδώ την κυρία Σόρενσεν. Είστε κάπου εδώ. Α, ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά είναι πάρα πολύ λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε τέτοια αμερόληπτη πληροφόρηση και μαρτυρίες για την πολιτική των θεωρήσεων. Για την ευρωπαϊκή πολιτική θεωρήσεων, τώρα μιλάμε για σύντομης διάρκειας θεωρήσεις βεβαίως. Και ήδη ακούσαμε ότι ίσως και να μην είναι το χειρότερο στον πλανήτη το σύστημά μας, είτε αυτό των θεωρήσεων είτε του Σέγγεν. Στις συστάσεις σας μιλάτε για ένα, ένα πλέγμα και ένα δίκτυο ε, συστάσεων και κανονισμών. Υπάρχει δηλαδή ο κανονισμό τη κάθε χώρα και μετά ο κώδικα των θεωρήσεων. Τι βασικού κανόνε πρέπει να εφαρμόζει κανεί για τι θεωρήσει και πώ να τι ε, εκδίδει. Αυτό θα αναθεωρηθεί. Είχαμε πρόσφατα δημόσιε διαβουλεύσει με κόσμο που ήρθε να μοιραστεί μαζί μα τι απόψει του για την πολιτική των θεωρήσεων Δεν συμμετείχαν όμως συγκεκριμένα ακτιβιστές ε, στις δημόσιες αυτέ διαβουλεύσεις στη μελέτη. Ε, οπότε δεν είχαμε σαφείς απαντήσεις. Αντί λοιπόν να τα λέμε μεταξύ μας, ίσως είναι η στιγμή να στραφούμε σε άλλους οργανισμούς ε, των κατών μελών. Πέραν των εργαλείων αυτών, έχουμε και τις συμφωνίες διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μεταξύ άλλων με το Αζερμπαϊτζάν, όπου η υποβολή κάποιων δικαιολογητικών είναι, πιο, είναι ε, απλουστευμένη και μετά έχει γίνει λόγος για έναν ορισμό, όντως, πράγμα δύσκολο. Δεν νομίζω ότι είναι... Δεν νομίζω ότι είναι μια γραμμή και ένας δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Προσπαθούμε όμως καθημερινά να ενισχύσουμε το δίκτυο συνεργασίας των κρατών μελών. Πολλέ φορέ έχουμε ιδιωτικέ εταιρείε, όχι οι κατοίκου φορεί των τρίτων χωρών. Ε, και φροντίζουν ως εκπρόσωποι να ε, διευκολύνουν τα πράγματα για τους ενδιαφερόμενους που δεν μπορούν να πάνε σε προξενείο αναγκαστικά ή πρεσβεία γιατί όλα αυτά συγκεντρώνονται συνήθως στις πρωτεύουσες των χωρών παίρνουν ένα μέτριο ποσό ως τέλος ε, τώρα δεν μπορώ να θίξω όλα τα σημεία των συστάσεών σας, οι οποίες είναι καλές, διότι λένε ότι υπάρχει κάποια βασική έλλειψη γνώσεων, αλλά ο κώδικας των θεωρήσεων έχει πρόσφατα αναθεωρηθεί. Έχουμε εξαλείψει τις ειδικέ κατηγορίες ετούντων. Για τον απλό λόγο ότι θέλουμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία έκδοση θεώρηση για όλου, όχι ειδικά για του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν σημαίνει ότι του χρειάζονται τι θεωρήσει πιο πολύ από άλλου εκείνοι. Έχουμε 60 εκατομμύρια αιτήσει ε, κάθε χρόνο. Όλοι έχουν θεμετού λόγου να αιτηθούν ε, θεώρηση. Πάντω υπάρχει ένα θεωρημένο κώδικα, ε, χωρί ειδικέ κατηγοριοποίησει, εκτό από του ναυτικού, αλλά εκεί είναι άλλη υπόθεση. Δεν θα περάσω σε αυτό το χωράφι έχουμε πιο γενναιοδόρο και ομοιογενές σύστημα έκδοσης θεωρήσεων με, την, με το σύστημα ντόμινο, για να το πω έτσι, δηλαδή εφόσον πάρει κανείς μια θεώρηση πρώτη φορά, μπορεί να φτάσει σε θεωρήση πενταετούς διάρκειας. Εδώ λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ελέγχει τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σέγγεν, βάσει του οποίου ε, βαθμολογούμε όλα τα κατημέλη στον τομέα του κεκτημένου του Σέγγεν και χρησιμοποιούμε και τις μελέτες ε, <clears throat> αξιολόγησης και αντικτύπου της Frontex και άλλων οργανισμών. Δεν καθόμαστε δηλαδή στα γραφεία μας και φανταζόμαστε τι έχει γίνει, αλλά πηγαίνουμε επί τόπου και συγκεντρώνουμε στοιχεία αποδεκτικά από γεγονότα και καταστάσεις. Αυτά εν γέννη. Ε, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ για αυτό που μας είπατε. Δείχνει ότι πρέπει να συζητούμε. Είστε ειδικοί στα θέματα θεωρήσεων, εμείς είμαστε ειδικοί στα ανθρώπινα δικαιώματα Νομίζω όμως ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να βοηθάμε και να προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν, ε, όσο αυξάνονται οι πιέσεις εναντίον τους, δεν πρέπει οι δικές μας υποχρεώσεις θεωρήσεων να τους δυσκολεύουν περαιτέρω τη ζωή. Δεν έχουμε χρόνο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει χρόνος για περαιτέρω συζήτηση με την Επιτροπή για το θέμα αυτό. Κάποιε παρανοήσεις σίγουρα μπορεί να λυθούν. Ευχαριστώ όλους σα τι προσκεκλημένου μα ιδίω και καλή τύχη και ευχαριστώ όλου σας. Είναι η τελευταία συνάντηση στην οποία προεδρεύω της ε, Επιτροπής σας. Ευχαριστώ όλους και θα επανέλθουμε. 13. Euh, Σημείο 13 της ημερησίας διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων για το τρίτο πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των δικαιωμάτων ανθρώπου και της δημοκρατίας. Έχουμε μαζί μας ε, την Λότε Κνούτσεν, ε, εκτελεστική διευθύντρια του Global Duandelom ε, από την, εξωτερική υπηρεσία, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Κιάρα Ντάμο, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Συνεργασίας της Κομισιόν και την Γκέιλ. Πώς να το πω αυτό το επώνυμό σας, ε, du sepulcre. Du sepulcre. Η κυρία Ντισεπίκλο λοιπόν από το δίκτυο Δικαιώματα Ανθρώπου και Δημοκρατία. Σημαντική είναι αυτή η στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη χτεσινή συζήτηση και την ακρόαση που είχαμε με τον κύριο Μπορέλ ε, για τη σχέση που έχουμε μεταξύ της δράσης του Κοινοβουλίου στα δικαιώματα του ανθρώπου και της δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης καθώς και την προετοιμασία του τρίτου προγράμματος δράσης. Η δουλειά που έχουμε ήδη κάνει είναι σημαντική. Ευχαριστώ την Ιζαμπέλ Βίσλερ στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου που έγινε για, το 2018 και που ήδη δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές συνενετικού χαρακτήρα στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δουλεύουμε πάνω σε αυτή τη βάση και πάνω στις διάφορες προτεραιότητες που έφεσε η υποεπιτροπή μας για το έργο που έχουμε αναλάβει. Όλοι ξέρουμε ότι ότι η εξωτερική πολιτική της Ένωσης θα αλλάξει από ένα πρόγραμμα δράσης. Αλλά αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα δράσης ως εργαλείο για να κατευθύνουμε τις φιλοδοξίες μας σε όλα όσα επιδιώκουμε για τη θέση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα στην πολιτική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου χωρίς να βλάψουμε άλλες πολιτικές εξωτερικές ή όχι. Το παράδειγμα προχθές που είδαμε στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δείχνει πόσο πρέπει να έχουμε συνέπεια στις θέσεις μας ε, στις εξωτερικές σχέσεις και πώς αντιλαμβάνονται οι εταίροι, οι χώρες εταίροι μας, έχουμε εταίρους σε όλο τον κόσμο, και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τα θέματα του δικαιω... των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο κέντρο των δράσεών μας. Δεν μιλώ για τη Σαουδική Αραβία, αλλά το ίδιο ισχύει και για το Ιράν. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε σε κάθε συνάντηση να θέτουμε το ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό όχι μόνο για τις εξωτερικές σχέσεις μας, αλλά και εσωτερικά, σε εσωτερικές πολιτικές ε, μέσα. Στον ευρωπαϊκό χώρο πρέπει να ακολουθούμε μια πολιτική δικαιωμάτων του ανθρώπου που θα σέβονται όλα τα κράτη-μέλη. Η δουλειά λοιπόν που κάνουμε, το έργο μας είναι ένα έργο πολιτικής συνοχής και πολιτικής συνέπειας. Και γι' αυτό και ένας λόγος για τον οποίο φέραμε εδώ την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι ακριβώς αυτός. Εμείς συνεργαζόμαστε με πολλές επιτροπές περιβάλλοντος, διεθνούς εμπορίου, με κάθε γενική διεύθυνση που έχει λιγότερο ή περισσότερο συνάφεια με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Προφανώς εμείς έχουμε έναν θεσμικό ρόλο, εσείς έχετε άλλο θεσμικό ρόλο, αλλά νομίζω ότι όλοι προς την ίδια κατεύθυνση πηγαίνουμε. Την οικουμενική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η έμφαση στην οικουμενικότητα των δικαιωμάτων είναι νομίζω καθοριστική σημασία. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην Λότε και κατόπιν στις υπόλοιπες ομιλήτρες και στα μέλη της Επιτροπής. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε, λέει η κυρία Κνούτσια να αναφέρει τον κύριο Μπορέλ. Και πρέπει να τονίσουμε ότι στο πρώτο του Συμβούλιο Εξωτερικών στις 9 Δεκεμβρίου στην Μέση Διατάξη είχε βάλει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αυτό δείχνει όπως είπατε ότι ο ύποδος εκπρόσωπος έχει δώσει προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι θέμα γεωπολιτικό. Ε, μέσα σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να θεωρούμε ότι είναι η σημαία αυτής της Επιτροπής και τη δεύτερη μόλις μέρα στη δουλειά ε, τότε που είχαμε εκείνο το φόρουμ των μη κυβερνητικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, έδωσε το μήνυμα πήγε ε, έκανε μια ομιλία και είπε ότι αυτό είναι από τα καινούργια θέματα που θα μας απασχολήσουν. Πρόκειται για την ε, πολυμερία της πολιτικής και φυσικά είναι αυτό ο σκοπός των δικαιώματα, αλλά είναι και θέμα πολυμερούς πολιτικής και οπότε αυτό είναι ένα συστατικό ε, αυτής της υπόθεσης, αυτούς της μεθόδου ε, εργασίας, αξιπολιτικής. Αν θέλει κανείς όμως να είναι ισχυρό και αποτελεσματικός, θα πρέπει να προωθεί συνέχεια, με συνέπεια τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα φόρα. Από τη Γενική Σύνδευση του ΟΗΕ, του Συμβούλου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ε, την Υπατιαρμοστία, όλα, παντού. Στο Συμβούλιο, Παντού, παντού θα πρέπει κανεί να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και εσεί ξέρετε περισσότερο από όλου ποια είναι τα προβλήματα σήμερα. Είναι σαφέ ότι υφίστανται τώρα πίεση, επίθεση. Μιλήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ω παγκόσμια αξία. Είναι ένα συστατικό τη ταυτότητά μα, τη ύπαρξή μα. αλλά ε, στη σημερινή συγκυρία αυτό δεν είναι αυτονόητο παντού σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι αξία δυτική και όχι παγκόσμια. Ε, είδαμε πολλά τελευταία που δεν τα είχαμε δει 70 χρόνια που πέρασαν από τότε που φτιάχτηκε ο χάρτης του ΟΗΕ. Είτε πρόκειται για επιθέσεις ακτιβιστές, είτε πρόκειται για πίσω γύρω στα δικαιώματα, εκμετάλλευση ανηλίκων, εργασία ανηλίκων, ε, παρεμβάσεις και επεμβάσεις ε, στην δημοκρατία, διώξεις κατά δημοσιογράφων. Άρα τώρα θα πρέπει να συσπηρωθούμε και να δώσουμε τη μάχη. Και έχουμε αυτή την ετησία έκθεση για την κατάσταση των δικαιωμάτων. Τώρα ήρθε την κατάλληλη στιγμή και βέβαια τα είπε έξω από τα δόντια ο κύριος Μπορέλη και είπε ότι θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο. Σας διαβεβαιώ η έκθεση θεωρούμε ότι συμβάλλει στο πρόγραμμα δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σήμερα συζητούμε. Είναι μια συμβολή σε αυτή την κοινή διαδρομή και ο χάρτης πορείας μας πρόκειται να βάλει τον πύχη της φιλοδοξίας ψηλά και θα μας απασχολήσουν όλα αυτά την επόμενη πέντα αιτία. Πρέπει να πούμε το πρόγραμμα δράσης έχει γίνει σημείο αναφοράς. Είναι μοναδικό στο είδος του. Παγκοσμίω. Μία πηξίδα. Είναι πλαίσιο αναφοράς για όλους τους εμπλεκόμενους. Κράτη, μη κρατικούς ε, παράγοντες παντού. Ε, για αυτό είναι σημαντικό να ανοίξουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο για αυτό το πρόγραμμα δράσης. Και με αυτό το πρόγραμμα δράσης έχουμε τις αξίες μας ως κοινωνία, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό διαπνέει όλο το πρόγραμμα δράσης και η ώρα είναι κρίσιμη διότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε για όλα αυτά τα προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε και το πρόγραμμα δράσης έρχεται τώρα σε ένα κομβικό σημείο και επίσης θα πρέπει να του δώσουμε μια νέα πνοή. Γιατί άλλαξε ο κόσμος. Ήρθε η ώρα να δούμε τις νέες προκλήσεις που αναδύονται. Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, ε, παραπληροφόρηση, δημοκρατία και αυτό πέραν όλων των βασικών αξιών μας. Θα πρέπει αυτά όλα να τονιστούν στο νέο πρόγραμμα δράσης. Έχουμε βέβαια και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το μέσο εξωτερικής πολιτικής, οπότε να εξασφαλίσουμε συνέπεια μεταξύ των πολιτικών μας είναι ευκαιρία να χαράξουμε την πορεία για την επόμενη πενταετία για να αντιμετωπίσουμε τα νέα προβλήματα. Είπαμε ότι θα εστιατούμε τώρα σε 5-6 σημεία, 5-6 κεφάλαια, πρώτα-πρώτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, χειραφέτηση, προστασία των προσώπων, ανθεκτικότητα, της ε, δημοκρατικής κοινωνίας, προώθηση ενός παγκοσμίου συστήματος για δικαιώματα και δημοκρατία ε, στα πλαίσια της πολυμερούς μεθόδου, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία και αυτά συνεργαζόμενοι. Τα ατομικά δικαιώματα βέβαια είναι στην καρδιά αυτής της διαδρομής, αποφύγη διακρίσεων, κάλυψη όλων των βασικών θεμελιωδών ελευθεριών με την υποχρέωση λογοδοσίας υπάρχει ένα κενό και έχουμε επίσης επιδείνωση σε σχέση με το κράτος του δικαίου και μας είπατε για την ε, συνοχή στην πολιτική μας και άρα θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τα κοινωνικά, δικαιώματα. Αυτά που τα προσέχουμε λένε και περισσότερο και τώρα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δράσης. Και έτσι βλέπουμε τι γίνεται τα διάφορα δικαιώματα, το δικαίωμα στο νερό, το δικαίωμα στην γη, όλα αυτά θα πρέπει να τα προωθήσουμε περισσότερο σε περισσότερα σημεία της υδρογείου. Επίσης και τα εργασιακά δικαιώματα και η σύνδεση με το εμπόριο και έχουμε το σύστημα γεμμένων προτιμήσεων συν και όλο αυτό το πλέγμα δικαιωμάτων βρίσκεται ψηλότερα σε σχέση με πριν στο θεματολόγιο της προτεραιότητας και η δημοκρατία όμως. Επίσης έχει αναδειχθεί επειδή βάσει των όσων προέκυψαν από τις εκλογέ παντού και έχουμε τις πιέσεις προς δημοσιογράφους, ελευθερία τύπου, ελευθερία λόγου ε, χρήση τεχνολογίας για να επηρεάσει κανείς εξελίξεις με παραπληροφόρηση, με πλατφόρμες, με την χειραγώγηση του, της κοινής γνώμης. Όλα αυτά εντάσσονται στις προσπαθίες μας και από πλευράς υπά του εκπροσώπου των δικαιωμάτων γιατί και εκείνος είναι και εκείνη είναι ε, αναφανδόν υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων και εκεί αποτελεί υψηλή προτεραιότητα το θέμα των δικαιωμάτων και το περιβάλλον. Να δούμε τι άλλο θα καλύψουμε σε αυτό το κομμάτι. Όλα αυτά είναι στα θεμέλια των προσπαθειών μας. Νέες τεχνολογίες και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί γιατί πάντα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τα θετικά της, ε, ε τεχνη, τεχνητής νοημοσύνης, ε, να εκμεταλλευτούμε τις εξελίξεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν κάποια ε, μείον, κάποια εκτήματα, είναι τα θέματα ηθικής για τα δικαιώματα και υπάρχει τώρα δανειτικό χαρτοφυλάκιο στην Επιτροπή Φοντερ Λάιεν. Οπότε γι' αυτό πάει στον εξωτερικό τομέα για να δούμε πώ θα προστατεύουμε το εκμεταλλευτικό με τον καλύτερο τρόπο χωρί να αποστερήσουμε του ε, ιδιώτε, τα άτομα από τα δικαιώματα και τι ελευθερίε. Ροή πληροφοριών, ε, προστασία ιδιωτικού βίου, προστασία δεδομένων. Αυτά, αυτά είναι επίση προτεραιότητα υψηλή. Αυτό απασχολούν τον ΟΗΕ στην Γενέβη, αλλά θα καλυφθούν και από την νομοθεσία. Για το πρόγραμμα δράσης και για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρέπει να δούμε και την κοινή γνώμη. Είναι κάτι που δεν πρέπει να μας ε, διαφεύγει. Είναι ένας επίσης σημαντικός χώρος. Πρέπει διαρκώς να συνδυάζουμε τις μερμηνέ μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τις συνδυάζουμε με τις παραβιάσεις που πραγματικά συμβαίνουν, αλλά να βλέπουμε και τα θετικά παραδείγματα. Έχουμε εντό αγγυλών αυτό που λέμε καλά παραδείγματα προ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θέλουμε να επικεντρωθούμε σε παραδείγματα από χώρε που έχουν φέρει αποτελέσματα. Μπορεί να είναι κάποιο νόμο, να είναι μια υπόθεση πρόσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακτιβιστέ πρέπει να δούμε τις εξατομικευμένες περιπτώσεις που έχουν πάει καλά. Μην ε, προκαλούμε κατάθλιψη μόνο και στενοχώρια σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Πρέπει αυτές τις υποθέσεις που βλέπουμε να τον κόσμο να τις γνωστοποιήσουμε. Πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμαστε Συνεργαζόμαστε μεταξύ μας οι συνάδελφοι που βλέπετε εδώ με τα θεσμικά όργανα, με τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνία των πολιτών. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι σημαντικό αυτό και βεβαίως με το Ευρωκοινοβούλιο. Είστε μέρος όλης, αναπόσπαστο όλης αυτής της διαδικασίας και υπό αυτήν την έννοια έχουμε επαφέ με μονομένε χώρε, με περιφερειακέ αρχέ που έχουν σημαντικό ρόλο. Εσεί προτείνετε λύσει ε, με την λογοδοσία που ασκείται. Η όλη συζήτηση για το τομέα αυτό πραγματικά μα παρέχει πολύτιμη στήριξη. Γι' αυτό λοιπόν ε, με τα χαράζει να ακούσω τα σχόλιά σας και βρισκόμαστε στη φάση όπου ελπίζαμε ότι θα είχαμε το πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο δεύτερο εξάμεινο, θα εξαρτηθεί και από την ε, κυλιόμενη ε, Προεδρία βέβαια, στο δεύτερο μάλλον 15 του Μαρτίου. Ευχαριστώ. Με αυτή την ημερομηνία κατά νου, πιστεύω ότι θα φροντίσουμε και εμείς κάτι να στείλουμε στον κύριο Μπορέλ νωρίτερα. Η κυρία Κιάρα Ανταμό τώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κνούτσεν έκανε μια πολύ συνοπτική επισκόπηση για τη δουλειά της ΕΕΒ και την ε, καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό μας ενδιαφέρει ακριβώς, η προετοιμασία του προγραμματος δράσης και αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχουν πέντε δις άνθρωποι που ζουν σε χώρες με δείκτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα να έχουν πολύ κακές επιδόσεις και αποτελέσματα. Τα πράγματα θα επιδεινωθούν και ξέρουμε ότι 111 χώρες τουλάχιστον βάσει των στοιχείων της κοινωνίας των πολιτών, 111 χώρες ανά τον κόσμο ασκούν πιέσεις στην κοινωνία των πολιτών, σοβαρές μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι ότι το όλο τοπίο και στο νέο αυτό πλαίσιο και στην αλλαγή του ε, πολυμερούς πλαισίου υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να ε, τα παίρνει τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά και να ε, διατρανώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε αυτό το τομέα και στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Ε, είναι λοιπόν ένα από τα εργαλεία αυτό που ετοιμάζεται για μας, το περιμένουμε πώς και πώς και για τη γεωπολιτική θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω θα μας τα, πούν, ε, μας τα είπε η κυρία Κνούτσεν και κυρία Ρενά, εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις βασικές ε, αξίες ε, στην καρδιά της δουλειάς της. Ε, αξίες και διαφάνεια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της Επιτροπής. Το πρόγραμμα δράσης για τη δημοκρατία πέραν αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό για το κράτος δικαίου, τα περιμένουμε. Και εξωτερικός, εκτός Ένωσης, πρέπει να δούμε το τι θέλουμε να πετύχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνίες δικαιοσύνης, ε, ευημερίας, βιώσιμες ε, χωρίς τα στοιχεία αυτά ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κάτω δικαίου. Είναι η ραχοκοκαλιά και για να πετύχουμε τις δεσμεύσεις μας βάσει της ατζέντα του 2030 και των στόχων της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, το 90% αυτών έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα τουλάχιστον από το 2016. Λέγονται μάλιστα SDG για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στα άλλα κεφάλαια των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, πάλι υπάρχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο τρόπος λοιπόν να επιτευχθούν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα δύο προτεραιότητα. Τώρα για την ε, σφαιρική προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Όπω είπε η κυρία Κνούτσεν, ίσω στο παρελθόν τα ζητήματα αυτά γίνονταν αντιληπτά ω ξεχωριστά μεταξύ του, δεν έβλεπαν τον άλλο σε σχετισμό. Τώρα έχουμε μια καλή ευκαιρία όμω αυτή η αλληλεξάρτηση ε, των τριών θεμάτων μεταξύ του να γίνει πιο σαφή. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα χωρί να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά ή να έχουμε ένα εύρυθμο δημοκρατικό σύστημα. Το πρόγραμμα δράση, ελπίζουμε λοιπόν, θα πάει σε αυτή την κατεύθυνση τη σφαιρική προσέγγιση. Δεύτερη παρατήρηση Θέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα αντιμετωπίσουμε με συνέπεια και στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτάζει την Πράσινη Συμφωνία και την εξωτερική της διάσταση. Είναι και αυτό μια σημαντική συμβολή. Να δούμε δηλαδή τις διασυνδέσεις περιβάλλοντος με ανθρώπινα δικαιώματα. Οι περιβαλλοντικές μέρημνες δεν πρέπει να πλήξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, του προσπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. η ψηφιοποίηση και η επίδρασή της στα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, την τεχνητή αυτή την αναφέρατε ήδη και μετά τρίτο ο προγραμματισμός. Πολύ σημαντικό για μα οι διαπραγματεύσει που έχετε για τα νέα εξωτερικά εργαλεία, το Ίνδικη, είναι ένα στρατηγικό στόχο να έχουμε μια προσέγγιση στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε όλα τα μέσα μας, όχι μόνο στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και μετά για το πρόγραμμα της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζουμε ότι μια ζωντανή, ζωηρή ε, και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών είναι σημαντικό. Ε, πρέπει όλες οι φωνές να μπορούν να ακούγονται και η αναπτυξική βοήθεια πρέπει να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών. Ιδάλω δεν θα χτυπήσουμε την ανισό, τις ανισότητες, ούτε θα πετύχουμε το στόχο της χιλιετίας ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν τις επιθέσεις των κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τις δούμε και από αυτή τη σκοπιά. Πραγματικά λοιπόν υποστηρίζουμε τη δουλειά που βρίσκεται υπό εξέλιξη στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δράσης. Θα είμαστε στη διάθεσή σας. Ίσως κάποιοι από εσά θέλετε πολύ λεπτημερείς δράσεις τώρα, οι οποίες να παρουσιαστούν, αλλά το εργαλείο αυτό πρέπει πρώτα να εκδοθεί και νομίζω ότι πιο σημαντικό από το το πρόγραμμα δράσης είναι ότι θα γίνει στην πράξη. Ευχαριστούμε κυρία Αδαμό. Η κυρία Ντουσεπίλ. Donc, Εγώ εκπροσωπώ μια μήκυο που ασχολείται και με ειδικά θέματα και με μια παγκόσμια προσέγγιση της ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου με συγκεκριμένες περιπτώσεις αγωνιστών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και εξετάζοντας την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ε, πολυμερούς προσέγγισης αυτόν τον καιρό. Η οργάνωσή μου είχε την ευκαιρία που να συμβάλλει μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στην επεξεργασία του σχεδίου δράσης. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, εδώ και εννέα μήνες. Η κοινωνία των πολιτών είχε την ευκαιρία να καταθέσει τις απόψεις της στην ΑΕΑ στο πλαίσιο μιας ε, γενικής διαβούλευσης που από ό,τι κατάλαβα δεν κάλυπτε μόνο την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και πήγαινε σε ένα ευρύτερο κοινό. Είχαμε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, πριν από δύο εβδομάδες για να λάβουμε το feedback ε, σε αυτά που είχαμε πει για την κατάσταση της επεξεργασίας αυτού του σχεδίου δράσης. Η διαδικασία διαβούλευσης οδήγησε σε κάποια απογοήτευση τους ε, μετέχοντες στο δίκτυο. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν αναγκαίο να προχωρήσουμε περαιτέρω στο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την επεξεργασία του προγράμματος με ουσιαστική αναγνώριση της θέσης και της σημασίας της κοινωνίας των πολιτών στην διαμόρφωση και διατήρηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής στο θέμα αυτό και στην αντιμετώπιση των επιθέσεων που δέχεται η κοινωνία των πολιτών για τα θέματα αυτά. Τώρα, πώς βλέπουμε τα πράγματα. με χαρά διαπιστώνουμε ότι κάποιες προτεραιότητες που προτείναμε έγιναν δεκτές στο πρόγραμμα δράσης. Έχουμε όμως και κάποιες ανησυχίες, ιδίως για την συγκεκριμένη διατύπωση, το wording που χρησιμοποιείται. Το πρόγραμμα δράσης έχει δεσμευθεί να προωθήσει τα δικαιώματα του ανθρώπου σε ένα εμπορικό πλαίσιο. Αυτή η διατύπωση δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε εμείς, ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να βοηθάει τα δικαιώματα των ανθρώπων επιτόπου. Σημαντικό είναι το θέμα αυτό, να υπάρχουν δηλαδή φιλόδοξες δεσμεύσεις και δυνατότητα συγκεκριμένης επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη βρίσκονται στην ίδια θέση με εμάς. Τι προτείνω λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε τους επόμενους μήνες για να έχουμε συγκεκριμένες συναντήσεις για συγκεκριμένα θέματα όπου θα μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε την εμπειρία που έχουμε για να περάσουμε από κάτι που είναι μια τυπικής ε, μορφής διαβούλευση και ενημέρωση σε κάτι που θα γίνεται περισσότερο ένας διάλογος ή μια εταιρική σχέση αν θέλουμε, με σαφείς καθορισμένους ρόλους ο καθένας. Ο καθένας έχει το δικό του χώρο, αλλά η κοινωνία των πολιτών έχει δύο πράγματα να προσφέρει. Πρώτον, εμπειρογνωμοσύνη. Δουλεύουμε με όλα τα θεσμικά όργανα. Ξέρουμε ότι κάποια μέλη της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης δεν έχουν συναντηθεί ποτέ με επιτρόπους, παρότι έχουμε να πούμε κάτι. Δουλεύουμε με όλες τις χώρες και επιτόπου. Έχουμε λοιπόν μια σφαιρική εικόνα. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν επιτόπου. Ξέρουμε τις δεσμεύσεις που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει όταν θέλει να πετύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο πλεονέκτημα που εμπλέκει την κοινωνία των πολιτών. Δεύτερο, η δυνατότητα αποδοχής των πολιτικών της Ένωσης. Αν έχουμε ευκαιρίες για να συζητήσουμε με τα θεσμικά όργανα, για να πρέπει να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος με παρουσίαση από όλες τις πλευρές των δικών τους θέσεων, κάτι που θα επιτρέψει και στην κοινωνία των πολιτών να μην το τορπιλήσει κείμενα που παρουσιάζονται πριν καν παρουσιαστούν. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η κοινωνία των πολιτών δεν είναι εδώ μόνο για να κατακρίνει, αλλά για να υποστηρίξει και να διευκρινίσει. Αυτά για το πλαίσιο. Ως προς το περιεχόμενο. έχουμε κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τις ε, ενημερωτικές συναντήσεις που μας δόθηκαν. Πρώτον, να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ συγκεκριμένων δράσεων και δράσεων αρχής. Προφανώς πρέπει να μείνει ευέλικτο το σχέδιο αυτό, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα, ιδίως για προτεραιότητες που δεν είναι πάντα εύκολες για μας. Στο πλαίσιο της ισορροπίας αυτής θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα που μας δημιουργούν τα σημαντικότερα προβλήματα. Επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών, επιθέσεις κατά της πολυμέρειας που σημαίνει παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα όλο και περισσότερο σε τομείς ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το ψηφιακό σύστημα και τις νέες τεχνολογίες. Για μας είναι σημαντικό το πρόγραμμα δράσης να προβλέπει δράσεις συγκεκριμένες με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας του διαλόγου, Δηλαδή, να περάσουμε από μια τυπική διαβούλευση σε μια πραγματική εταιρική σχέση, να δίνουμε έμφαση στην προστασία των αγωνιστών. Δεν μπορεί να έχουμε καλές πολιτικές αν δεν, πολιτικές αν δεν έχουμε και κάποιους αγωνιστές για τα δικαιώματα των ανθρώπων που είναι επιτόπου και μπορούμε να προστατεύσουμε. υπάρχουν πολιτικές και συστάσεις που θα, μπορέσουμε, που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε πιο ολοκληρωμένα. Για παράδειγμα, οι συστάσεις της Συνόδου του Παρισιού του 18 για τους αγωνιστές. Τώρα, αγωνιστές και κοινωνία των πολιτών. Το θέμα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι πρόκληση προς τα έξω, αλλά είναι πρόκληση και προς τα μέσα. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτρέψουμε στην κοινωνία των πολιτών να έχει ευέλικτα ευέλικτους πόρους που θα της επιτρέψουν να κάνει δράση όχι μόνο με λίγα άτομα και reporting αλλά και να αντιδρά ουσιαστικά στις επιθέσεις κατά των αγωνιστών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για το θέμα της πολυμέρειας. Εγώ θεωρώ σημαντικά ότι η πολυμέρεια, η πολυμερής προσέγγιση δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να χρησιμεύει για την βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων του, του ανθρώπου. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες δράσεις, μπορεί να γίνει, να κάνει περισσότερα η Ένωση σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα. Για παράδειγμα, η Ένωση έχει την τάση να χρησιμοποιεί το item 5 του διαλόγου στα πλαίσια του ΙΕ για τα αντίπεινα για να υπογραμμίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις και χώρες. Είναι σημαντικό να το δούμε στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής προστασίας των δικαιώματων ανθρώπου της Ένωσης. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε δράσεις που ασκούνται κατ' εφαρμογή των guideline μαζί με, το, με την πολυμερή προσέγγιση για να ενισχύσουμε το ρόλο του ΟΗΕ στα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα πρέπει να θέσουμε και το ζήτημα του membership, της συμμετοχής. Ε, κράτη που είναι γνωστά για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που χρησιμοποιούν την πολυμερή προσέγγιση για να μειώσουν την οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δημιουργούν, συνιστούν ένα πρόβλημα. Άρα, η λύση περνάει από το να υποβάλει η Ένωση περισσότερες υποψηφιότητες από αυτές που έχει δικαίωμα. Δεν γίνεται αυτό τώρα. εταιρική σχέση με τον κλάδο, όλοι οι, όλα τα μέλη του, της πλατφόρμας ε, τονίζουν την ανησυχία τους για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορεί να εμπλέκει το ιδιωτικό τομέα χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και κάθε μέρα βλέπουμε καταπάτηση των δικαιωμάτων ε, ε, ακόμα και από την Ευρώπη και σε πολλές περιπτώσεις όπως σας έχουμε πει δεν θέλω τώρα να σας τα πω αλλά είναι πολύ σημαντικό πολύ σημαντικό ε, πρόκειται για αυτό το, την κατευθυντήρια αρχή και αυτόν έχει συνέπεια με τη δράση της Ένωσης σε όλα τα φόρα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ναι είμαι υπέρ της εφαρμογής διεθνώς αυτών των αρχών του ΟΗΕ ναι, αλλά όμως τι γίνεται, γιατί δεν τα λέγει στον δυτικό τομέα αυτό είναι πρόβλημα να και μια συγκεκριμένη πράξη για τα ψηφιακά τώρα ε, έχουμε πάρα πολλά στο πρόγραμμα δράσης για την ψηφιακή τεχνολογία πολύ σημαντικό για το μέλλον θα, και οπότε θα πρέπει να προπαρασκευαστούμε δύο τινά. Πρώτα πρώτα η κοινωνία θα πρέπει να αναπτύξει τις δυνατότητες. Πολύ σημαντικό αυτό να καλυφθεί από το πρόγραμμα δράσης. Οπότε επομένω περισσότερη πόρη περισσότερο capacity building, περισσότερη συνεργασία με την ε, κοινωνία. Και έτσι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι έτσι αναβαθμίζονται οι δυνατότητες της κοινωνίας για να ανταποκριθεί και δεύτερον ε, για τα ψηφιακά θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερος κάτι. Κάτι το οποίο τώρα προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η προβληματική, οι κοινωνικές πλατφόρμες σε σχέση με την μετάδοση των πληροφοριών προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί γιατί ε, για την παραπληροφόρηση ακριβώς μετράνε αυτές οι κοινωνικές πλατφόρμες και άρα θα πρέπει να καταπολεμηθεί κάθε επίθεση κατά της δημοκρατίας. Να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι κοινωνικές πλατφόρμες αυτό κάνουν. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για κάποιες εικόνες, εικόνες από το Ισλαμικό κράτος και άρα καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οπότε θα πρέπει και μέσω του ιδιωτικού τομέα να δούμε πώς λειτουργεί μια τέτοια επιλογή των φωτογραφιών που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και αυτό είναι κατά της ε, ελευθερίας ε, έκφρασης, ε, κατά των ακτιβιστών, οπότε έτσι θα πρέπει να δημοσιεύονται κάποια πράγματα τα οποία είναι βλαπτικά για αυτές τις αξίες μας. Επομένως θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την υπεραπληροφόρηση ε, όσον αφορά κάποια ξενά κράτη τα οποία ε, μεταδίδουν τέτοιε πληροφορίες οπότε γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι πλατφόρμες ε, θα πρέπει να τους δώσουμε την δυνατότητα της επιλογής αλλά έχουν αποκτήσει κάποια ισχύ. Η δε ποιότητα της πληροφορίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μείνει υπό τον έλεγχο του δημοσίου και κάποιες εγγύσεις προς τους ακτιβιστές. Ε, αυτό κάνει ο φορέας μας. Ε, έχουμε αυτή την έκθεση με τον Ντουτέρντε στις Φιλιππίνες που είναι, πώς να το πω έτσι διπλωματικά, ε, αγενής μέσω του Facebook. Και αυτό δεν έχει χειραγώγηση, είναι ένα γεγονός. Οπότε αυτό ε, μεταδίδεται. Και το θέμα είναι για το Facebook κατά πόσο να πούμε ε, τα πρέπει να ανέβουν, πρέπει να δημοσιοποιηθούν στην χιλή. Να, όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε, να δούμε τα όρια της δύναμης των ε, κοινωνικών πλατφόρμων. Τώρα, όσον αφορά τις αρχές για το πρόγραμμα δράσης, είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε το πρόγραμμα δράσης κάποιες ε, γενικές ε, πρωτοβουλίες που υπάγονται όμως στις ε, αρχές μας, το αδιέρετο των δικαιωμάτων, το παγκόσμιο, η συνέπεια στην πολιτική. Θεωρώ ότι είναι προβληματικό ότι υπάρχουν κάποιες δραστηριότητε για να προωθήσουν στο εξωτερικό τα δικαιώματα χωρίς να βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των πολιτικών της Ένωσης γιατί πολλές φορές υπάρχει μια διαρκής επίδραση στον κόσμο και άρα θα πρέπει να δούμε με ποιους μηχανούς, μηχανισμούς μπορούμε αυτά να τα εποπτεύσουμε και να τα επιδιορθώσουμε το ΣΥΠΗΝ. Άρα είναι θέμα αξιοπιστίας της Ένωσης στο εξωτερικό, της συνέπειας ε, όσον αφορά την προσήλωση στη συνθήκη ε, και να δούμε με τι δραστηριότητες μπορούμε να προωθήσουμε αυτές τις αρχές στα τρίτα κράτη, αλλά να προσέξουμε τις δικές μας δραστηριότητες. Οπότε και το τελευταίο για τις αρχές που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε τις δράσεις για τα ίδια τα μέσα πολιτικής της Ένωσης. Πολύ ωραία, ναι, να καθορίζουμε και τις προτεραιότητες. Το θέμα είναι όμως το πού θα ενεργήσουμε, που θα δράσουμε, αλλά να έχουμε τα απαραίτητα αποτελεσματικά μέσα προς τούτο. Και γι' αυτό και εγώ στέκομαι σε τρία μέσα πολιτική. τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διάλογο για τα δικαιώματα και το πώ θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη αλληλεπίδραση των διαφορετικών μέσων πολιτικής. Αυτά τα τρία θα πρέπει να πλησιωθούν με τι δράσει. Και για να κλείσω το θέμα της εποπτείας, της παρακολούθησης, όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε, θέλουμε εταιρική σχέση με την κοινωνία. Θέλουμε να συγκροτηθεί task force, έτσι να έμπλακουν όλοι οι ενεχόμενοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βούλιο, η κοινωνία, τα κρατη αλλά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή και να την προσαρμόσουμε, προσαρμόσουμε το πρόγραμμα ε, όποτε υπάρχει κάποια έκθεση σχετικά λένε ότι υπάρχει αιτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την εξωτερική, από την εξωτερικής δράσης και ότι αυτό αρκεί όχι γιατί όχι δεν μπορεί να είναι απλή αξιολόγηση η παρακολούθηση, η πλαισίωση του προγράμματος δράσης. Α, πρέπει να έχουμε κριτική ματιά για να μπορέσουμε να δούμε αν πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μπορεί αυτό να στριμώχνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζεται αυτός ο έλεγχο αυτή η εποπτεία. Άρα μπορεί να χρειαστεί ομάδα εργασία για αυτό το λόγο. Ευχαριστούμε Γκαέλ για αυτή την τόσο περίπλοκη, εξαιρετικά περίπλοκη παρουσίαση. Νομίζω ότι όλοι, οι τα θεσμικά όργανα έχουν κάθε λόγο να θέλουν να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών. Είναι επικοδομητικό αυτό. Ε, και οι συστάσει σου ήταν ε, πολύ σκόπιμε. Θα συμφωνήσω και με τη ΛΟΤ. Και εδώ Πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση επικοδομητική για να αξιοποιήσουμε ό,τι έχει γίνει σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Θετικέ κινήσει που επιτρέψαν στα θεσμικά όργανα για ορισμένα θέματα να προχωρήσουν ακριβώ γιατί συνεργάστηκαν και στηρίχθηκαν στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου. Βλέπω ότι η Ζαμπέλ Βισλέρ έχει ζητήσει το λόγο, η Λίντα και φαντάζομαι και η Άννα. να ευχαριστήσω τις τρεις ομιλήτρες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας ακούει κανείς. Je voudrais euh, revenir sur différents éléments que euh, Madame Κάποια από τα στοιχεία που ανέφερε η κυρία Sepulcre. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρατε, ότι όλοι έχουμε τα δικά μας όρια και ότι πρέπει να κοιτάζουμε τους περιορισμούς του καθενός. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι το λέτε. Διότι πραγματικά αυτό που μας νοιάζει είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό μπορεί να κάνει η κοινωνία των πολιτών. Και αυτό που καταγγέλει η κοινωνία των πολιτών δεν γίνεται το ίδιο με τον ίδιο τρόπο από τι αρχέ. Δεν, μπορεί, δεν μπορούν οι αρχέ να καταγγείλουν, να καταγράψουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και τόσο ευθέω. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση, έχουμε τον ίδιο σκοπό. Δεν συμφωνούμε πάντοτε για το ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε και να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και να θέλαμε. Είναι αυτό μια πολύ καλή βάση όμως για να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας. Γιατί πραγματικά πρέπει να βάλουμε τα σωστά ε, θεμέλια για την ε, αποτελεσματικότητα. Το είπαμε και προηγουμένως. Είπαμε ένα μητρό για τους υπερασπιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το συμπέρασμα είναι ότι πιο επικίνδυνο θα ήταν κάτι τέτοιο και πιο δύσκολο να εφαρμοστεί και μάλλον αντιπαραγωγικό. Αυτό για να επισημάνω, να πω τη δουλειά που γίνεται είναι συνήθως πολύ πιο περίπλοκη και ε, πολύ πιο διεξοδική από αυτό που βλέπουμε στην επιφάνεια. Και έπειτα να πω ότι μιλάμε πολύ. Στο κοινοβούλιο λέμε πολλά, πολλά ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ίδιο. Εμείς ζητάμε πολλά πράγματα, προφορικός, γραπτός και επανειλημμένος. Και να επιμείνω στο εξή γιατί είναι σημαντικό για τους περισσότερους από εμά, ιδίω σε αυτή τη χρονική φάση, γιατί μας απασχόλησε από καιρό. Έχουμε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ. Θέλουμε ένα μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό το ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το οργανώσει. Είναι μια συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ισχύει και γενικότερα. Όταν πραγματικά θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα, δεν αρκεί να μιλάμε και να αγορεύουμε μόνο ή να ζητάμε απλώ τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται και από πράξει. Πρέπει να υπάρξει κάπου και μία υλοποίηση όσων λέγονται. Θα ήθελα να πάψω σε αυτό, διότι ήθελα ακριβώ εκεί να επιμείνω. Ο μηχανισμό παρακολούθηση είναι το πιο σημαντικό και θέλω αυτό να συγκρατήσετε από όλη μου την παρέμβαση. Πραγματικά εκτιμώ πολύ τη δουλειά σα. Πρόεδρο, ευχαριστώ Ιζαμπέλ. Επειδή ξεπεράσαμε κατά κάποιο, κατά το χρόνο μα, για τη Διερμηνία μας μένουν τα γαλλικά και τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα πρωτογαλλικά. Οι συντονιστές είναι ήδη εδώ. Απλώς ε, για τους διερμηνείς θα εργαστούμε με τις γλώσσες των συντονιστών προβλέποντας στις 11. Ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας πρωινό.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 And without those flexibilities, including the possibility to work with unregistered partners, the possibility to work without consent of the government, a lot of the actions we are talking about here today would not simply be possible. Thank you. Oui, je voudrais juste réagir sur la question du commerce et combien la DG Trade est maintenant impliquée pour défendre les droits de l'homme. Je voudrais quand même souligner que